Good morning, colleagues. Can we start? Please to be... Συνάδελφοι, καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Just missing five meters for Gunnar. Welcome. So let me open today's uh, econ Λοιπόν, ας ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε δύο εκθέσεις ε, και κάποιες ψηφοφορίες και μετά άλλη μια έκθεση. Οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου είναι πάρα πολύ σύντομες. Να έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης ε, φαντάζομαι εγκρίνεται. Δεν έχω κάποια άλλη ανακοίνωση. Και τίποτα να σας πω για τις δύο οργανικές ε, διαπραγματεύσεις ε, της προηγούμενης εβδομάδας. Παίρναμε λοιπόν στο σημείο 4. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016, όπως ξέρετε είναι παραδοσιακή έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας επί της έκθεσης της ΕΚΤ για να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις ε, και την απάντηση της ΕΚΤ και υπάρχει έτσι η δυνατότητα άσκησης δημοκρατικού ελέγχου. Έχουμε λοιπόν τον Γιώνας Φερνάντες και τους σκιώδες ηγητές. Πέντε λεπτά εισηγητής, τρία λεπτά οι σκιώδες ηγητές και δύο λεπτά για την διαδικασία του Catch the Eye. Τον λόγο λοιπόν έχει ο συνάδελφος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, σήμερα σας υποβάλλω εδώ στην Επιτροπή την ετήσια έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου της διαχείρισης του κεντρικού ε, ευρωπαϊκού άμπου για με ένα βασικό μήνυμα, ότι δεν είναι καιρός τώρα να τροποποιήσουμε το βασικό μας μήνυμα. Καταρχάς διότι με όλα τα μέτρα θέλουμε να επιδιώξουμε τις ε, τον επανέλθει ο πληθωρισμός στο 1%. Το προηγούμενο χρόνο ήμασταν στο 0,2%. Ε, όμως ε, οι προβλέψεις για φέτος τοποθετούν στο 1,5% τον πληθωρισμό, στο 1,3% για το 2018 και στο 1,6% για το 2019. Οπότε η Ευρωζώνη θα μπορούσε να διανύσει 7 ε, χρόνια ε, πολύ, μακρύ, πολύ μακριά από τον στόχο. Βρισκόμαστε σε μια αποπληθωριστική φάση. Αυτό το θεωρούμε θεωρούμε θετικό, αλλά ακόμα είμαστε πολύ μακριά από την επίτευξη του στόχου, όπως είπα. Δεύτερον, είναι σαφές ότι η οικονομία φαίνεται να έχει μπει σε μία φάση ανάπτυξης χάρη στην νομισματική πολιτική και την εξέλιξη των, ενεργειακών, των τιμών ενέργειας. Εν τω μεταξύ έχουμε μηδενική ε, δημοσιονομική όθηση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δε θετικούς, ε, θετικά ποσοστά, ενώ σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είμαστε στο 1,2% για το 2016 και θα παραμείνουμε σε αρνητικά ποσοστά τουλάχιστον για δύο ακόμα χρήσεις. Άρα η Ευρωζώνη προσφέρει μη πληθωριστικές ε, ευκαιρίες σε ένα χρονικό ε, διάστημα ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ΑΕΠ μας ε, αλλά χωρίς να πιεστούν οι τιμές το ενεργό, η ενεργή ανάπτυξη για τα επόμενα τρίμηνα και για τα επόμενα χρόνια θα παραμείνουν σε μια ε, περίοδο μη πληθωριστική. Ε, στην έκθεση που υποβάλλουμε σήμερα εκτεμούμε, αξιολογούμε μάλλον τα διάφορα ε, ομόλογα με την χρηματοδότηση με νέου είδους πιστώσεις. Θεωρούμε πως όλα αυτά είναι θετικά, αν και ζητούμε περισσότερη διαφάνεια όχι μόνο για την χρηματοδότηση που δίνεται, αλλά και για τα κριτήρια της επιλεξιμότητας ε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για τις μικρομεσαίες, ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο συμφωνούν με το πλαίσιο της Συμφωνία του Παρισίου. Θέλουμε να επικρατήσει ένα ομοιογενές πλαίσιο για όλες τις χώρες και ιδιαίτερα για τη δημοκρατία της Ελλάδας, μια χώρα που χρειάζεται την αλληλεγγύη μας για να μπορεί να παραμείνει και στην Ευρωζώνη. Όσον δε αφορά την οικονομική μας πολιτική, η χώρες ε, θα πρέπει να παραμείνουν στο 5% ε, ανάπτυξη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μέλλον ε, και να μπορέσουμε φιλόδοξα να εφαρμόσουμε την νομισματική μας πολιτική. Υπερασπιζόμαστε τις θετικέ επιπτώσεις των μέτρων μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την περιορισμό των πτωχεύσεων. Θέλουμε να παραμείνουμε δραστήριοι όσον αφορά την ε, δυνατότητα να κατανομής χάρη στην νομισματική πολιτική, καθώς και τη συμβολή που μπορεί αυτή να έχει στον περιορισμό του πληθωρισμού, ώστε να έχουμε ε, πραγματικά έσοδα. Η έκθεση επίσης ε, απηχεί την Τραπεζική Ένωση και την προώθηση αυτής για να μπορέσουμε έτσι να ολοκληρώσουμε το γενικότερο πρότυπο. Όσον αφορά το μέλλον της Ευρωζώνης, ε, θέλουμε να έχουμε ένα ελεύθερο ενεργητικό για, ε, ε, για να μπορέσουμε να δράσουμε, αλλά και να μπορέσουμε να έχουμε τα ωφέλη που θέλουμε για τον προϋπολογισμό της Ένωσης χρειάζεται να συζητηθεί μια μεταρρύθμιση και το, η Επιτροπή των, του Προϋπολογισμού έχει πρόσφατα υποβάλει μια τέτοια αναφορά όσον αφορά αυτή μου την άποψη την οποία επαναλαμβάνω. Όσον αφορά το Brexit, δεν θα πρέπει να μείνουμε στις παραδοσιακές μας ε, θέσεις. Αυτή η έκθεση αποτελεί μια βάση για συζήτηση. Είναι ανοιχτή στην συζήτηση και στις, ε, σε τροπολογίες. Θα θέλαμε να έχουμε μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση για να μπορέσουμε να την εγκρίνουμε τους επόμενους μήνες, έτσι συνεισφέροντας τη βελτίωση της νομισματικής πολιτικής και του ελέγχου αυτής που καθημερινά γίνεται και επηρεάζει την καθημερινή ζωή ε, χιλιάδων πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Ο Σίγκφιτ Μούρεσαν ε, είναι σκιώδης εισηγητής ε, για το ΕΛΚ, αλλά από ό,τι κατάλαβα ο Μπούλχαρ Πάλς ε, θα μιλήσει στη θέση του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ ο Σίγκριτ Μουρεσάν δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Θα ήθελα όμω εκ μέρου του να ευχαριστήσω τον εισηγητή Γιώνα Φερνάντε για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμή. Το σχέδιο έκθεσης αποτελεί καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις ανάμεσα στον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Ο Σίγκφριντ Μούρεσαν θεωρεί σημαντικέ τι εξή τρει προτεραιότητε για την έκθεση που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Καταρχά, τον πρωταρχικό στόχο του ΕΛΚ, όπω καθορίζεται στι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τρίτον, μεταρρυθμίσει στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καταρχάς, ε, λοιπόν, ε, ο βασικός στόχος ε, της νομισματικής πολιτικής είναι να διατηρηθεί η σταθερότητα των τιμών που καθορίζεται με στόχο για, την, για τον πληθωρισμό κοντά αλλά κάτω από το 2%. και όχι 2% όπως αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητος οργανισμός και η ανεξαρτησία του είναι απαραίτητη για να μπορεί να πετύχει το βασικό του στόχο, την σταθερότητα των τιμών. Δεύτερον, επικροτούμε τον ε, διάλογο για νομισματικά θέματα που ε, διασφαλίζει την ε, λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινό. Και τρίτον, ο πρόεδρος Μάριο Τράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν χάνει ευκαιρία να τονίσει τη σημασία των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα του, στην ζώνη του ευρώ. Και όπως έχει πει, η νομισματική πολιτική από μόνη δεν μπορεί να κινητοποιήσει την οικονομία εάν δεν συμπληρώνεται από ε, δημοσιονομικές πολιτικές ε, και μεταρρυθμίσεις ε, για αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητα στα κράτη-μέλη. Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστούν ευνοϊκές συνθήκες για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος πρόθεση των ε, επενδύσεων για να ε, έχουμε ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Ε, όπως έχει πετύχει επιτυχώς ε, η Επιτροπή μας ε, στην έκθεση του 2015, θα πρέπει πάλι να στοχεύσουμε η ε, έκθεση αυτή να επικεντρώνεται στα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να αποφύγουμε τις συζητήσεις για αρμοδιότητες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, περιμένουμε την έκθεση για ε, την Τραπεζική Ένωση και θα πρέπει να στείλουμε σαφές μήνυμα από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016. Αυτές λοιπόν είναι οι προτεραιότητες του Σίγκφριτ Μοριζάν για την έκθεση και προσβλέπει στη συνέχιση των συζητήσεων στις επόμενες συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών και θα ήθελα να ευχαριστήσει και πάλι τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ευχαριστή. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Μπουρκχάρτ. Νομίζω ότι ήσουν άξιος αντικαταστάτης. Τον κύριο Λούμες από το ECR, αλλά αν κατάλαβα καλά, θα μιλήσει ο κύριος Λούκα εκ μέρους του. Εγώ θα εκπροσωπήσω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ τον συγητή για την έκθεση του, την οποία θεωρώ ως μια αφετηρία για την συζήτηση η οποία βεβαίως παρουσιάζει τη σοσιαλδημοκρατική άποψη, κάτι το οποίο εντάξει είναι λογικό αλλά δεν μπορεί να βρει την σύμφωνη γνώμη του ECR. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να σας υποστηρίξω. Μιλάτε για τον όγκο του CSPP ο οποίος θα πρέπει να δημοσιευτεί και το ίδιο βεβαίως και για τα επιχειρηματικά δάνεια. Σας υποστηρίζω στην κατεύθυνση της ε, διαφάνειας. Αλλά βεβαίω ε, μετά ακολουθούν διάφορα πράγματα που δεν έχουν ούτε μία σχέση με την κεντρική τράπεζα. Π.χ. αυτά τα οποία λέτε για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να αντισταθμιστούν τα υπερβολικά πλεονάσματα. Αυτό δεν, είναι, δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά και την εντολή της Κεντρικής ε, Τράπεζας. Επιπλέον Βεβαίω, όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα πάντα έχουμε κατά νου την Γερμανία, αλλά η Γερμανία με την Ευρωζώνη έχει έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον είναι λογικό να μιλήσουμε για μείωση του υφιστάμενου πλεονάσματος μιας χώρας. Επίσης, η απέτηση για την κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηριχθεί από την Κεντρική Τράπεζα και αυτό είναι εκτός της εντολής της ε, τράπεζας. Επίσης, ούτε μία σχέση δεν έχει με η απέτηση για τα European Safe Assets, δηλαδή ένα άλλο όνομα για τα ευρωομόλογα. Και αυτό δεν είναι δουλειά της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, δεν έχει εντολή να στηρίξει την Ελλάδα. Η εντολή της Κεντρικής Τράπεζας είναι η σταθερότητα των τιμών και όχι η στήριξη της Ελλάδας οι απαιτήσει να στηριχθούν οι βρετανικές εκείνες ε, τράπεζες οι οποίες θέλουν να φύγουν από τη Μεγάλη Βρετανία και να έρθουν στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν είναι δουλειά της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης δεν ήταν μέλος της Ευρωζώνης ποτέ η Μεγάλη Βρετανία. Οπότε τι δουλειά έχει εδώ πέρα η ε, Κεντρική Τράπεζα. Επίσης η απέτηση τα κέρδη της, ε, το λεγόμενο σένιορας να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραβιάζει τις συνθήκες και την εντολή της Κεντρικής Τράπεζας. Η απέτηση μιας χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής ε, και η αγορά κρατικών ε, ομολόγων αλλά ακόμα και δανειοδότησης βεβαίως ε, δεν έχει ούτε μία σχέση με την εντολή της χιλιοδρικής όπως και το PSPP και τα άλλα σχετικά προγράμματα επίσης αντιβαίνουν στο δίκαιο καθώς πρόκειται η κρατική ε, νομισματική χρηματοδότηση. Επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες πτυχές που λέτε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση για τα αποτελέσματα των stress test και ακολούθησε η κατάρρευση των ε, Ισπανικών ε, και Ιταλικών τραπεζών ενώ είχαν περάσει τα τεστ. Αυτό είναι σωστό. Επίσης η τράπεζα πλέον δεν έχει κάποια δυνατότητα για να διορθώσει την ανατίμηση του ευρώ, ούτε αυτό το έχετε αναφέρει και επίσης η ποσοτική χαλάρωση εκρεμεί ενώπιον του ε, ευρωπαϊκού δικαστηρίου μετά από μια προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο που παρέπεμψε το θέμα εκεί. Επίσης, μιλάτε για τον υπολογισμό του ΑΕΠ και για το πώς βεβαίως θα πρέπει να στοχεύει το ονομαστικό ΑΕΠ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά αυτό, όπως λέτε και εσείς αλλού, πάλι δεν είναι δουλειά της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, τώρα έχουμε τους ε, ομιλητές από το Άλντερ. Ε, κύριος Τρεμόζα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ζουμπόφσκι που είναι κανονικά ο σκιώδης για αυτή την έκθεση λείπει και γι' αυτό θα σας αναφέρω κάποιες δικές του παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες για το σχέδιο έκθεσή σας. Ε, πολύ πλήρης έκθεση που θα ανοίξει την συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στους σκιώδεις. Εν γέννη, ε, βλέπει θετικά την έκθεση αυτή, αλλά θέλει να τονίσει ότι μια έκθεση ε, σε ομα, ε, τέτοια θα πρέπει να είναι περιορισμένη και περιεκτική. 39 παράγραφοι ωστόσο υπάρχουν εδώ, ίσως να υπάρχει μια τάση για μια μακριά έτσι, έκθεση, μακροσκελή έκθεση, ενώ εκείνος προτιμά να μείνουμε στα όσα είναι αρμοδιότητες της μονομισματικής πολιτικής και όχι να μπούμε σε άλλα θέματα. Επίσης ε, πιστεύει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, αλλά θέλει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλές από τις ενέργειες ε, αυτές που προβλέπονται δεν θα λειτουργήσουν χωρίς ε, συμπληρωματικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Οπότε οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στην νομισματική πολιτική για να λύσουν τα ε, μόνιμα διορθωτικά τους προβλήματα. Αυτή είναι μια θέση που η ομάδα μου συμμερίζεται και ήθελα να αντιλάβετε υπόψη. Τέλος, μια άλλη παρατήρηση, η παράγραφη 7 και 8 της έκθεσής σας, όπου κάνετε λόγο για Δηλαδή για χρήματα που φέρνει ένα ελικόπτερο ξαφνικά ε, θα πρέπει ίσως να το συζητήσουμε περισσότερο ε, μεταξύ των σκιωδών αλλά και μιλώντας για στόχο, στόχοθέτηση ονομαστικού ΑΕΠ θα είναι κάτι δύσκολο να δεχτούν πολλά από τα μέλη της ομάδας μας. Τέλος, μια συμβουλή τα τελευταία χρόνια η έχει καταφέρει να έχει μεγάλη συνένεση στην Ολομέλεια. Γύρω στο 80% των μελών υπερψήφισαν. Εδώ βέβαια η έκθεση αυτή δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι σημαντική εάν το Κοινοβούλιο φτάσει σε ε, πλειοψηφία και μάλιστα μεγάλη πλειοψηφία. Στο παρελθόν είχαμε σημαντικές βελτιώσεις για τα θέματα διαφάνειας, για παράδειγμα. Το 2012 είχαμε την η δημοσίευση των ισοζυγίων και το 2014 είχαμε επίσης διαφάνεια για τις αγορές CSPB. Μάλλον αυτό έγινε πριν από κάποιους μήνες. Πήραμε τα ονόματα και πληροφορίες, μερικές πληροφορίες, όχι πλήρης. Οπότε είναι καλύτερο κατά τη γνώμη της ομάδας μου να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία παρά να έχουμε μόνο μια ιδεολογική νίκη για κάποιες θέσεις που όμως στην ουσία θα είναι ήττα για το Κοινοβούλιο και θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την εκτεκτός ε, αυτού του σώματος. Ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε την άποψη της ομάδας σας και τώρα έχουμε τον, τον εκπρόσωπο της ΓΚΟΕ, τον κύριο Παπαδημούλη. Δεν είναι εδώ, οπότε έχουμε έναν αντικαταστάτη του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρου ε, του κυρίου Παπαδημούλη που δεν ε, μπορεί να είναι παρόν για τη συζήτηση αυτή και θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει ε, στο όνομα του αν συμφωνείτε. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση τη οικονομική και νομισματικής πολιτική. Δυστυχώ, οι λύσει που παρέχουν οι οργανισμοί όπω είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αρκούν για να λυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και ω μέλη τη επιτροπή μα. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορε πτυχέ του ρόλου που παίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η έκθεση των ε, τραπεζικών συστημάτων ε, σε κρίσεις ε, και προβλήματα ρευστότητας, καθώς και η επιμονή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες, αποτελούν δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό εντός της Επιτροπής μας. Επίσης, τις πολιτικές που θα μπορούσαν να είναι θετικέ για κάποιε οικονομίε, όπω είναι η ποσοτική χαλάρωση, δεν σχεδιάστηκαν σωστά και δεν εφαρμόστηκαν εγκαίρω. Η αμέλεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, στο τομέα αυτό οδήγησε σε αύξηση τιμών σε πολλές περιπτώσεις. Η ε, έλλειψη δυναμικού εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, σημαίνει ότι συνταξιοδοτικά ταμεία απαντούν προβλήματα και γι' αυτό αυτό επιβαρύνει ε, τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να συζητηθεί. Υπάρχουν λοιπόν ανησυχίες και για τις πιο ασθενείς οικονομίες της ζώνης του ευρώ αλλά και για το ενιαίο νόμισμα στο σύνολό τους. Θα πρέπει λοιπόν να συζητηθεί και το μείγμα πολιτικής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και ο ίδιος ο θεσμός. Θα πρέπει να έχουμε ένα πιο δημοκρατικό μοντέλο, διότι το ε, δημοκρατικό έλλειμμα χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να ασκείται πίεση σε οικονομίες των κρατών μελών και να λαμβάνονται αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει τις ε, αποφάσεις του ε, θα πρέπει να υπάρξει νομικό καθεστώς για τους κατακέλλοντες παρατυπίες εντός ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς ε, κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και μάλιστα πολύ σωστά στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν δεν έχουν μόνο να κάνουν με τους κανόνες ε, και τους κανονισμούς, ε, οι μεταρρυθμίσεις ε, θα πρέπει να αφορούν την όλη τη δομή για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί σε οδό ανάπτυξης. Στο όνομα του κ. Παπαδομήλου θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον εισηγητή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις πάνω στην έκθεση αυτή σε επόμενες Σας ευχαριστώ κατόπιν για τους πράσινους Μουριν Σκοτ, η ίδια. Ναι, ναι, και εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Ζητώ συγγνώμη. Και εγώ να ευχαριστήσω τον συγγητή. έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ πέρα. Μια πάρα πολύ καλή έκθεση που ελαμβάνει πολλά σημαντικά ζητήματα. Ιδιαίτερα χαιρόμαστε που βλέπουμε την πρόταση στην παράγραφο 8 που ζητάει η έκτενα να συνδέσει στόχο τη σταθερότητα των τιμών με την ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ. Επίση, χαιρόμαστε για την πρόταση στην παράγραφο 7 που λέει ότι θα πρέπει να σχετεί μια επέκταση του προγράμματο Τέλτρο στα νοικοκυριά μέσω δανείων μηδενικού επιτοκίου. Θεωρούμε ότι έτσι θα έπρεπε να διοχετευτούν οι πόροι των τραπεζών προς αηφόρες δραστηριότητες. Όπως ξέρει ο συγητής, το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών φαίνεται ότι έχει επιτύχει να κινητοποιήσει την ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά και θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τη σταδιακή κατάργησή του. Όμως ε, χαίρομαι που υπάρχει ακριβώς ε, το ζήτημα της ε, στρέβλωση τη αγορά Θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τους Ευρωπαίου πολίτες. Βεβαίω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για την ΕΚ την οποία επιβάλαμε. Εμείς, η Επιτροπή μας Οραμών και η επιστολή που υπογράψαμε και βεβαίως καλωσορίζουμε την απόφαση της ΕΚΤ να αποκαλύψει ποια εταιρικά ομόλογα έχει αγοράσει. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη διαφάνεια και να αποκαλυφθούν όλα τα εταιρικά ομόλογα. Πλέον θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής των εταιριών για να μην συγκρούεται με άλλους στόχους της ε, τράπεζας. Επίσης, ίσως η άρνηση ακριβώς μιας ε, πλήρους απάντησης σε αυτό το θέμα οφείλεται σε έναν φόβο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το πώς θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις. Είχαμε παραδείγματο χάρη μετοχέ τη ΣΕΛ, το ΤΑΛ, ΡΕΠΣΟΛ κτλ. Θα συμφωνήσουν νομίζω οι βουλευτέ μαζί μου για το ότι υπάρχει μια παράκαμψη των κανόνων τη ε, Τραπεζική Ένωση ε, στην περίπτωση τη ε, Ιταλία. και θα πρέπει ακριβώ να δούμε πόσο κοινοβούλιο θα πρέπει να μην υπάρξει κάποια υπονόμευση του ρυθμιστικού πλαισίου και εισαγωγή ενός στοιχείου ηθικού κινδύνου. Τέλος, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προγραμματίζει τις ε, μελλοντικέ της σχέσεις ε, με το City του Λονδίνου όταν θα γίνει τρίτη χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βεβαίως ε, δεν ξέρω το τι θα σημαίνει αυτό για τα φορολογικά έσοδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει στόχος να διατηρηθεί ο ενίο χαρακτήρα τη ενία αγορά. Και θα πρέπει να έχουμε μια πιο ξεκαθαρή ιδέα για το πώ θα γίνει μια τέτοια ρύθμιση και τι θα γίνει σε περίπτωση αποτυχία των διαπραγματεύσεων και ενό άτακτου Brexit. Σα ευχαριστώ. Για το EFTD Μάρκο Βάλλη. σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ που μπορούμε να συζητήσουμε ή θα βάλουμε τροπολογίε γραπτό για κάποια σημεία σε σχέση με παλιότερε εκθέσει, είναι ένα βήμα μπροστά. Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, είναι απαράδεκτο που δεν τονίζεται με αποφασιστικό τρόπο η πραγματικότητα της Ευρωζώνης ε, και κατά συνέπεια και τον, τα αποτελέσματα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι μια κεντρική τράπεζα που σήμερα δεν μπορούμε παρά να ε, παρανασκήσει η πολιτική ε, ε, υπάρχει μια πολιτική κόντρα ανάμεσα στις χώρες ε, που, δεν μπορούν πια να, να υιοθετήσουν πιο αδύναμο ε, νόμισμα. Πρέπει να γίνει αναφορά όσον αφορά την έλλειψη ισορροπίας, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος, ποια, προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να συνεχίσουμε. Να να έχουμε αυτό το, αυτό το νόμισμα ή να περάσουμε σε μια επόμενη φάση όπου θα έχουμε ε, πολιτική, νομισματική, όχι μόνο ευρωπαϊκή, αλλά παγκόσμια, που θα οδηγεί στην ανάπτυξη της χώρας, όταν θα έχουμε δηλαδή μια ε, επόμενη φάση όπου τα παλιά προβλήματα του ευρώ θα συνεχιστούν ε, και θα έχουμε ακόμα πιο έντονη κρίση, αν δεν τα λύσουμε τώρα. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να τονιστούν περισσότερο αυτές οι δυσκολίες και αν δεν το κάνουμε, οι συνέπειε θα είναι πολύ σοβαρέ και από πολιτική άποψη θα έχουμε χάσει μεγάλη ευκαιρία, γιατί θα έχουμε μόνο αντιπαρατευθεί σε άσχετα θέματα, ενώ στην πραγματικότητα το, βασικό πρόβλημα είναι ότι μία νομισματική πολιτική δεν μπορεί να καταλήψει 19 διαφορετικές απαιτήσει όσον αφορά επιτόκια και πληθωρισμό. Και εκεί είναι ε, το σημείο κίνησης για κάθε ουσιαστική συζήτηση. Έχουμε και σημαντικές ε, διαφορές ε, για τη Τραπεζική Ένωση. Και εδώ θα υποβάλουμε τροπολογίες με τις υπόψεις μας όσον αφορά κάποια στοιχεία που οδηγούν σε έλλειψη ισορροπίας. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Στη διάρκεια των συζητήσεων με τους σκιώδεις, στις διαδοχικέ συζητήσει θα υποβάλω και αυτές τι απόψει. Και επίση είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η νομισματική πολιτική σήμερα είναι και πάντα ε, όλο και λιγότερο επηρεάζει την πραγματική οικονομία. Αν δούμε την ανεργία, ε, τους ε, ανθρώπους που είναι αδρανείς, αλλά και τα στοιχεία για την πραγματική οικονομία, θα δούμε πως είναι πολύ πιο ψηλά από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, ειδικά στις περιφερειακές χώρες. Άρα λοιπόν αυτή η νομισματική πολιτική πώς θα γίνει να επηρεάσει την πραγματική οικονομία. Μήπως υπάρχει κίνδυνος φούσκας πάλι. Αυτός είναι κίνδυνος ο μεγάλος και πρέπει να προσέξουμε να μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία. Οι νομισματικές πολιτικές λοιπόν πρέπει να δούμε αν είναι ε, ε, αποτελεσματικές ή είναι ένα φάρμακο που το δίνουμε ε, και πολλές φορές τελείως ανεύθυνα. Να εμβαθύνουμε, να εμβαθύνουμε πολιτικά, αλλά με όλους τους συναδέλφους, γιατί φαίνεται να είναι σταθερή η κατάσταση σήμερα, όμως σε λίγο καιρό θα έχουμε ένα πρόβλημα με μια φάση καθοδική στην οικονομικό κύκλο και πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ε, τελευταίος είναι ο κύριος Άνεμανς από το ΙΕΝΕΦ. E Τρία λεπτά. Και εγώ ε, θα μιλήσω ε, για μένα. Μια έκθεση αυτή έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Λέει ότι ε, πρέπει να μην ασχολείται καθόλου με το νόμισμα η Κεντρική Τράπεζα. Προσπερνά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεπεράσει την έντολη της η Κεντρική Τράπεζα, κατά το οποίο βεβαίως δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο στην Καλσρούη. Και η ποσοτική χαλάρωση, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεπεράσει την εντολή της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας. Η οικονομική πολιτική είναι αρμοδιότητα κατά κύριο λόγο των κρατών μελών και σύμφωνα με το δικαστήριο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται το ζήτημα νομισματικό αλλά είναι ένα θέμα οικονομικής πολιτικής. Αυτά αναφέρει όπως σας λέω ε, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι σημαντικοί λόγοι φαίνεται ότι δείχνουν ότι υπάρχει εδώ πέρα μια υπέρβαση της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία σε αρχιτές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Βεβαίως αυτά θα έπρεπε να τα λάβει υπόψη και η κυρία Μέρκελ η οποία το 2013 έκανε μια πολιτική συμφωνία με Ιταλία και Γαλλία για την χρηματοδότηση της ε, Ελλάδος, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μην υπάρχει καμία διάσωση και καμία χρηματοδότηση κρατών. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, δεν υπάρχει πλέον ακριβώς η πολιτική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία ήταν η Λιδία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος ε, και θα πρέπει να αναλυφθεί δράση και να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντός του πλαισίου της εντολής της. Και δεν μπορούμε άρα να στηρίξουμε αυτή την έκθεση γιατί απέχει από την πραγματικότητα και ξεπερνάει πολύ απλά το γεγονό ότι η έκτεχη ξεφύγει από την εντολή της πλέον την έχει θυσιάσει στον βωμό μιας νομισματικής ένωσης η οποία ήταν βασισμένη σε ένα λάθος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, έχουμε άλλους ομιλητές, ούτε χρόνο έχουμε. Να δώσω δύο λεπτά στον Ιώνα αν θέλει να κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια και για τις ε, από αποτιμήσεις των συναδέλφων σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα περιμένω με ανυπομονησία όλες τις τροπολογίες που θέλουν να υποβάλουν για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και ε, όσον αφορά τα όσα είπε ο συνάδελφος Ραμόνα της Άλντε, τελευταία έχουμε μεγάλες ε, συμφωνίες ε, όσον αφορά την ΕΚΤ και ελπίζω πως μετά από τη συζήτηση και τις διαπραγματεύσεις και σε αυτή την περίπτωση θα πάμε σε μια συνένεση ευρεία από πλευράς αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον κύριο Τσαμπών που θέλει δύο λεπτά για το Catch the έτσι θα έχουμε κρυπήσει το χρόνο μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να υποβάλω στον ε, Χωνάς που έκανε τεράστιο έργο και στους υπόλοιπους που δουλεύουν ε, για αυτό το θέμα μία παρατήρηση πώς ακριβώς βοηθήσουμε στο να εστιάσουμε καλύτερα τα προβλήματα. Ε, το, πρόβλημα είναι, ε, το πρώτο θέμα είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και αυτό δεν θα γίνει και δεν θα έχουμε τραπεζική ένωση παρά μόνο όταν αυτό το σύστημα θα υπάρξει. Πού είναι λοιπόν αυτή η αλυσίδα προθεσμιών, ας πούμε, αυτή η αλληλουχία των προθεσμιών για να μπορέσει αυτό να θεσπιστεί εφόσον όλοι υποτίθεται το θέλουμε. Πιστεύω πως είναι ρόλος αυτού του Κοινοβουλίου να άρει τα πολιτικά εμπόδια για να έχουμε την συνείδησή μας ήσυχη ότι το προσπαθήσαμε. Πιστεύω πως, αυτό το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων είναι ουσιώδες για να μπορέσουμε να έχουμε τραπεζική ένωση, γιατί διαφορετικά κατά τη γνώμη μου δεν θα το καταφέρουμε. Όσο ευρωπαϊστής και να είναι κανείς, δεν πιστεύω πως θα υπάρξει ε, τραπεζική ένωση χωρίς αυτό. Αυτό το σύστημα εγγύησεων έχει ήδη, έχει ήδη εγκριθεί. Οπότε θέλουμε ένα σχέδιο ε, εγκαθίδρυσης το οποίο να δίνει βεβαιότητα στις αγορές. Γιατί διαφορετικά ε, θα φτάσουμε σε το δεύτερο σημείο το οποίο επίσης θέλω να ζητήσω από τα μέλη της ομάδας να εγκύψουν σε αυτό και να προβληματιστούν γιατί παρακολουθούμε μια, ένα περιορισμό της ε, Τραπεζικής ε, Ένωσης γιατί όλες οι διεθνείς δραστηριότητες των τραπεζών, όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, όλη η ε, ευρωπαϊκοποίηση της Ένωσης, της Τραπεζικής Ένωσης πάει πίσω και έχουν χαθεί 3 εκατομμύρια ευρώ. Ε, τράπεζες γερμανικές ε, ε, επανεθνικοποιούνται, επανεθνικοποιείται η τραπεζική πρακτική και θα πρέπει να μας απασχολήσει το γιατί. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Κλείσαμε λοιπόν το θέμα αυτό. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 13 Σεπτεμβρίου, εξέταση τροπολογιών 9-10 Οκτωβρίου, ψηφοφορία 20-21 Νοεμβρίου στην ΕΚΟΝ και δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πότε θα πάει στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για αυτήν την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Δεν είχαμε ακριβώ συνένεση, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και προχωράμε στο σημείο 5 που είναι η δική μας ε, γνωμοδότηση για την έκθεση ΛΥΜΠΕ για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει πολλά μέτρα, έχει εγκρίνει διάφορα νομοθετήματα για το θέμα αυτό. Ε, γνωρίζετε ότι η δέσμευση ε, κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Συντάκτης της νομοδότησης μας είναι ο Φούλιο Μαρτουσιέλο και του δίνουμε 7 λεπτά για την εισαγωγή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε δίκιο. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, ε, πολύ θεμελιώδες για να αποφύγουμε το να μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει το έγκλημα. Με αυτή τη διάταξη αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αποφύγουμε το να είναι αποδοτικό το έγκλημα. Θέλω να σας υποβάλω λοιπόν αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για ένα θέμα τόσο σημαντικό και για το οποίο είμαι εισηγητής. Το θεματικό πλαίσιο επί το οποίο θα εργαστούμε αναπτύσσεται με ενδιαφέροντες τρόπους ε, γιατί στόχο έχει την δέσμευση κερδών που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Η δέσμευση των αγαθών εγκληματικών οργανώσεων είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπος για να μειωθούν οι εγκληματικές δυνατότητες τους και για να περιοριστεί η ταχύτητα ανάκαμψή τους. Γιατί αυτό πλήττει αυτά που για αυτούς είναι το καύσιμο, δηλαδή το χρήμα. Αυτό μας ε, βοηθά να καταλάβουμε πόσο είναι απαραίτητη μία πλήρης διάταξη, ένα πλήρες νομοθέτημα, ώστε να μπορεί να ασκηθεί, να υπάρξει προστασία ε, και ένα είδος αντιπαράθεσης στο οργανωμένο έγκλημα. Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπόλ που παρατίθεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι παράνομες αγορές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδουν 110 δις ευρώ που προέρχονται από εγκλήματα και το 98% αυτών παραμένει στα χέρια των εγκληματιών. Είναι μια τεράστια, ε, μια τεράστια όγκος χρημάτων που επανεπενδύονται σε εγκληματικές δραστηριότητες και γι' αυτό ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι να δουλέψουμε με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να βελτιώσουμε τη δομή ώστε να είναι σε θέση να δεσμεύσει, να παγώσει και να δημεύσει αυτά τα αγαθά. Ε, συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικά καθεστώτα ανάκτησης, δέσμευσης. Αυτό είναι προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικής σημασίας και όπως επιβεβαιώνει και η Κομισιόν θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση ε, καταδικών και δικαστικών αποφάσεων. Και αυτό είναι σημαντικό κλειδί στο πλαίσιο της ασφάλειας. Προχωρώντας τώρα στην ανάλυση των ισχύων των, ε, των, ισχύων των κανόνων, ε, των μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης, τα μέτρα εναρμόνισης ε, με τις ρυθμίσεις πλαίσιο και την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ιδέα είναι να διευρυνθεί το πλαίσιο παρέμβασης, να ξεπεραστούν τα όρια που μπορεί να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά του, γιατί η ουσιαστική έννοια της ε, δικαιοσύνης ε, εδράζεται στην ε, συνεργασία στο ποινικό και στο αστικό δίκαιο. Και έτσι θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος σε ένα σύστημα που θα αναγνωρίζει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα νομικά συστήματα άλλων χωρών τις δικαιοδοσίες άλλων χωρών ως έγκυρες και αναγνωρίσιμες χωρίς να χρειάζονται άλλες διατυπώσεις. Όπως διευκρινίζεται και από το κείμενο που έχουμε υποβάλει, η συνεργασία, η διασυνοριακή είναι απαραίτητη απολύτως ανάμεσα στα ποινικά, ε, ποινική δικαιοσύνη και τις υπόλοιπες ε, αρμόδιες εθνικές αρχές και είναι ουσιαστική για τη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος της Ένωσης καθώς και για την ε, αξιοπιστία του. Η αρχική πρόταση λοιπόν, όπως συντάχθηκε, στόχο έχει να διευρύνει τον νομοθετικό πλαίσιο ε, και να επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση και την ε, δυνατότητα εκτέλεσης των διατάξεων περί δέσμευσης. Ε, Με αμοιβαία αναγνώριση λοιπόν ποινικών αποφάσεων. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην αρχή ο κανονισμός αυτός να μπορεί να εφαρμοστεί σε, για όλες τις διατάξεις κατάσχεσης που ε, διατάσσει μια δικαστική αρχή ή αρμόδια ε, αρχή. Ε, τροπολογία 3 Πρέπει δηλαδή να προβλέπουμε τη δυνατότητα δέσμευσης μετά από μία διαδικασία, μία ποινική διαδικασία, ποινική δίωξη ή λόγω αστικής, ε, μάλλον απόφασης αστικού δικαίου. 50% ε, του ποσού με την εκτέλεση της διαδικασίας δέσμευσης θα πρέπει να μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης της απόφασης, χωρίς να, ε, τον κανόνα που προβλέπει αυτό να συμβαίνει τη στιγμή που τα ποσά που έχουν δεσμευθεί είναι ίσα με ή, μεγαλύτερα από τα 10.000 ευρώ. Και αυτό ως αποζημίωση των κρατών για τις δραστηριότητε τις οποίες έχουν προβεί, τις ενέργειες που έχουν προβεί. Ε, συχνά υπάρχουν ε, και διάφορες δαπάνες για τη διαχείριση όλων αυτών, ενώ η δραστηριότητε οι διασυνοριακέ μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε διάφορε χώρε, η ποινική διαδικασία και η δικαστική διαδικασία που οδηγεί στη δέσμευση γίνεται μόνο σε μία χώρα. Άρα λοιπόν τα. Ε, ε, χρήματα από τη δέσμευση πρέπει να απο... πηγαίνουν στην εκδόσα αρχή ώστε να καλυφθούν τα σχετικά έξοδα και σχετικές δαπάνες. Η Κομισιόν λέει επίσης ότι το σημερινό σύστημα δυστυχώ δεν λειτουργεί. Έχει διαπιστωθεί ότι τα κέρδη από διακίνηση ναρκωτικών δεν μπορούν να κατασχεθούν ούτε να δεσμευθούν λόγω της έλλειψης διασυνοριακής συνεργασίας σε επίπεδο ε, δικαστικών αρχών. Και γνωρίζουμε δυστυχώς ότι η διακίνηση ναρκωτικών είναι ένα μέσο που όλες οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτήσουν τις διάφορες τους δραστηριότητες. Είναι λοιπόν προφανές Περιμένω ε, την συμβολή των συναδέλφων ώστε μαζί να εργαστούμε για αυτό το θέμα. Thank you very much. Uh, Shadow for is... Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Εύανα από το S&D, ο συζητητής. Παρακαλώ, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Συμφωνούμε πλήρως με το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εθνικές αρχές να οδηγήσουν τους ένοχους στην δικαιοσύνη και πρέπει να ανακτηθούν οι απώλειες ε, και βεβαίως να δεσμεύονται τα προϊόντα εγκλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δρανοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια και να επεκταθεί το δίκτυο και άλλο πέρα από το ρευστό. Και βεβαίως καλωσορίζουμε τα θέματα φορολογικής απάτης, ε, χειραγωγήσεις ε, της αγοράς, ε, των συμβάσεων και βεβαίω τους διάφορους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επενδυτικών ταμείων. Και επίσης το άρθρο 3 θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή για τα τρία έτη ποινή φυλάξης. θα πρέπει να μιλήσουμε για το ότι κάποιες χώρες εκτός της Ένωσης διασφαλίζουν ε, την ανωνυμία των διεφθαρμένων ανθρώπων που στέλνουν λεφτά εκεί πρέπει λοιπόν να δούμε το τι γίνεται με τις ε, τρίτες χώρες ε, και τη μεταφορά κονδυλίων εκτός Ένωσης και μετά να υπάρχει αυτή η προστασία και η ανωνυμία. Πρέπει να σκεφτούμε και την διπλωματική οδό. Θα τα πούμε αυτά βεβαίως ε, και στους κοιόδης Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε την κυρία την Ευχαριστώ. πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτουσέλο για το σχέδιο έκθεσής του. Εξετάζοντα τις δεύτερες διαφορετικές ε, γνωμοδοτήσεις που υποβλήθηκαν, ε, βλέπω ότι ο εισηγητή ε, Λίνς επέλεξε την επιλογή Β που σημαίνει ότι ε, η δέσμευση και δίμευση ε, και για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή ε, αυτού του κανονισμού. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε οι κανόνες αυτοί να παραμένουν συμβατοί με την νομοθεσία των κρατών μελών. Δεν συμφωνώ με όλε τι προτάσει του εισηγητή, ε, πιστεύω όμω ότι θα πρέπει να συζητηθούν όλε οι πιθανέ λύσει. Κάποιε από τι τροπολογίε έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη των χρηματοπιστωτικών αγορών ε, και επικεντρώνονται ιδιαίτερα στι καταχρήσει στον τομέα αυτών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή γιατί ε, επικεντρώνεται ειδικά στο θέμα αυτό. Ποιο είναι το συγκεκριμένο θέμα που θέλετε να λύσετε και γιατί δεν καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία η διαχείριση ε, και διάθεση των ε, δεσμευμένων περιουσιακών ε, στοιχείων θέλετε να χωρίζονται εξίσου ανάμεσα στο κράτος μέλος αίτησης και εκτέλεσης εφόσον βρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο κατόφλι. Θα ήθελα όμως να ακούσω γιατί αυτός ο καταμερισμός κατά 50-50% και ε, θα ήθελα να ακούσω επίσης αν υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Σας ευχαριστώ για την εκθεσή αυτή και προσβλέπω στι στις περαιτέρω συζητήσεις μας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να ελέγξω μόνο αν υπάρχει κάποιος εδώ από το ECR. Δεν είναι κανείς παρόν. Ε, πράσινη. Εύα Ζολή. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, τον κύριο Μαρτουσέλο. Συμφωνώ απολύτως με την ε, πρόταση και επιθυμία για ρύθμιση στον τομέα αυτών ε, και την αμοιβή αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Στο παρελθόν υπερβολικά ποσά έχουν εξατμιστεί μόνο και μόνο λόγω της διαδικασίας που εφαρμοζόταν στο πλαίσιο της απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου που δεν λειτουργούσε καλά. Συμφωνούμε λοιπόν στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου. Επίσης, συμφωνούμε να καλύπτεται όχι μόνο ο ποινικό τομέα, ε, αλλά και οι διοικητικέ διαδικασίε. Συμφωνούμε δηλαδή με το ευρύ πεδίο εφαρμογή αυτή τη ε, έκθεση και μπορείτε να ε, βασίζεστε στην υποστήριξή μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω την Μπάρμπα Κάπελ, κανέναν άλλο από το ΙΕΝΕΦ. E ε, μας μένουν λίγα λεπτά για τη διαδικασία Catch the Eye. Υπάρχει κανεί που να θέλει να πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανεί. Ε, να ξαναδώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Μαρτουσέλο για να κλείσει τη συζήτησή μας. E ευχαριστώ πάρα πολύ τους εισηγητές ε, που παρενέβησαν γιατί βεβαίως όλα αυτά θα συνεισφέρουν στο να εμπλουτίσουμε την πρόταση, να τελειοποιήσουμε το κείμενο και να το μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε στον στόχο που είναι η δέσμευση των προϊόντων εγκλήματος. και να μην έχουν έτσι ακριβώ ε, τα μέσα για να κάνουν άλλα εγκλήματα. Έχουμε λοιπόν τα θέματα τα οποία είπαμε, την αμοιβαία αναγνώριση, τα ποσοστά και τα σχετικά και είναι προφανές ότι μιλάμε για μια μεγάλη πρόκληση ότι πρέπει να προετοιμάσουμε μια έκθεση στην οποία η κατάσχεση θα είναι αποτελεσματική και θα είναι έτσι ε, κάτι το οποίο θα αποτρέπει από την διάπραξη εγκλημάτων. Αυτά και ευχαριστώ τους συναδέλφους για αυτή την πρώτη ανταλλαγή ιδεών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε... Ναι, εδώ ολοκληρώνω τη συζήτησή μας. Να σας υπενθυμίσω τον χρόνο. Έχουμε 12 Σεπτεμβρίου τη καταστροπολογιών, εξέτασή τους 9 και 10 Οκτωβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 6 Νοεμβρίου. Ξέρουμε πώς μιλάμε για γνωμοδότηση για την ΛΥΜΠΕ μόνο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα διακόπτουμε για 15 λεπτά και θα επανέλθουμε για την ε, ψηφοφορία στις 6 παρατέταρτο. Ευχαριστώ.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 online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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Ε, θα παρακαλούσα πρώτα να κάνουμε μια δοκιμή. Παρακαλώ τοποθετήστε την κάρτα στο μηχάνημα και κάνουμε δοκιμαστική ψηφοφορία. One ένα vote. Άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Ωραία, κλείνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε από το σχέδιο γνωμοδότηση τη Μόλι Κοτκέιτο για ε, όσου αποκαλύπτουν εμπιστευτικέ πληροφορίε. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε έναρξη της ψηφοφορίας. APP discussing. Το ΕΛΚ συζητάει. Okay. Can I close the vote? Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35, υπέρ. Κατά. Αποχές. S&D. Πρέπει να ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά δεν είδα τα χέρια σας. Έναξη της ψηφοφορίας, τροπολογία 35. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβιβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Έλεγχος έναρξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση, έναξη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση, έναρξη της ψηφοφορίας. Άλλοι δύο συνάδελφοι να ψηφίσουν. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αυτή ήταν η J. Συμβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρι... εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 81, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 81, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 85, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική A, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική B, Β, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 8, έναρξη της ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 15. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 36 υπέρ, Κανείς δεν καταψήφισε, 13 αποχές, εγκρίνεται η έκθεση, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Προχωράμε τώρα στο περίσεμα από την ε, προηγούμενη ψηφοφορία που είχαμε, που είναι το δεύτερο τμήμα της ε, γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό. Η είναι ο Μάρκους, συντάκτης είναι ο Μάρκους Φέρμπερ. Θα θυμάστε ότι πρόκειται για το τμήμα που ε, Ε, περιέχει τον σχολιασμό. Ήδη έχουν ε, ψηφιστεί ε, οι γραμμέ του προπολογισμού. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β, Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 21, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβιβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ή, e, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53, υπέρ, κατά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 Παρακαλώ, θα ήθελα απλά να εκφράσω την ανησυχία μου. Ε, με εκπλήσει που ε, ψηφίστηκε με τόσο ευρία πλειοψηφία η ε, γνωμοδότηση του Μάρκους Φέρμπερ που μήπως έχει χάσει ε, την ακμή του μετά από τόσα χρόνια στο Κοινοβούλιο Πρόεδρος, όπως βλέπετε είχαμε θετικές εξελίξεις ε, τα τελευταία, ε, τις τελευταίες μέρες ε, και είχαμε νέες συμβαστικές τροπολογίες. Ε, και όπως βλέπετε εξελίσσεται ο Μάρκος. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα είχα πλειοψηφία. Παραγίνεται καλός ο Μάρκος. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για το σχέδιο γνωμοδότησης της Μαρίας Αματίας για την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης. Πρόκειται για γνωμοδότηση για έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης. Σας παρακαλώ να σοπάσετε. Έχουμε λοιπόν έκθεση της Επιτροπής απασχόλησης και εξετάζουμε τώρα τις τροπολογίες. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Παρακαλώ, Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Ehm, Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν τους διάφορους συναδέλφους, ε, ε, σκιώδεις εισηγητές. Βεβαίως μιλάμε για μια γνωμοδότηση που έχει ως θέμα το θέμα των, της ανισότητας, πολύ ευρύ θέμα που αγγίζει πολιτικές, οικονομικές αλλά και κοινωνικές πολιτικές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της, ανά... της εξέτασης αυτής της έκθεσης ε, κατάλαβα ότι δεν θα πρέπει μόνο να βάλουμε την, ε, να φτιάξουμε μια γνωμοδότηση, αλλά να ε, μιλήσουμε και για όλους τους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας, αλλά να προσπαθήσουμε να ε, εστιάσουμε περισσότερο το κείμενο με τα δικά μας θέματα. Ευχαριστώ λοιπόν για τις τροπολογίες και με αυτή την προτασή θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύνολο από διάφορες ε, παραγράφους που ε, αρχικά είχαμε περιορίσει γιατί ε, περιοριζόμαστε από τις διατάξεις που ισχύουν για το μέγεθος των γνωμοδοτήσεων και βασικά θέλω να σας συνοψίσω τις γραμμές στις οποίες κινούνται αυτές οι νέες παράγραφοι με βάση τις συμβολές των συναδέλφων. Θα πρέπει να δείτε ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, τροπολογίες που δεν ε, έχουν συμπεριληφθεί στη συμβιβαστική λύση ε, μάλλον ε, σε συμβαστικές τροπολογίες. Οι προ, συμβαστικές προτάσεις λοιπόν που σας ε, έστειλα και που θα ήθελα να έχω τα σχόλιά σας έχουν σχέση με την εισαγωγή παραγράφων για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η αύξηση των ανισοτήτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Μια άλλη προσέγγιση έχει να κάνει με την ανάγκη δημόσιων και ιδιωτικών καταθέσεων ως στοιχείο κλειδί στην καταπολέμηση των ε, ανισοτήτων και στην ε, ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μια τρίτη γραμμή είναι να φτιάξουμε μια νέα συμβιβαστική πρόταση για την παιδεία και την ε, επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα των ε, δημοσιονομικών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των νέων τεχνολογιών Έχουμε να κάνουμε λοιπόν εδώ με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον πολιτιστικό αποκλεισμό. Έπειτα, οικονομικές πολιτικές δικαιότερες από αυτές που περιλάμβανε η αρχική πρόταση, πιο δίκαιες, πιο αποτελεσματικές και γι' αυτό και εκτιμώ τις συμβολές ε, και τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα προς φορολογικούς παραδείσους, ε, αλλά και την αποφυγή του ΦΠΑ και προσπαθώ μάλλον να φτιάξω και μια ε, κοινή πρόταση με βάση αυτές τις τροπολογίες για να τις συμπεριλάβω στην τελική έκθεση. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε ένα μέσο ε, και να χρησιμοποιήσουμε την ανισότητα, τις κοινωνικές πολιτικές και την ανεργία ως έναν από τους ε, δείκτες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα εθνικά προγράμματα, της μεταρρυθμίσεις και αυτό έγινε με βάση τη συμβολή των διαφόρων ε, συναδέλφων και της τροπολογίας τους. Ελπίζω να σας ακούσω σε σχέση με αυτές τις προτάσεις που έλαβαν και να επιβεβαιώσω ακόμη μια φορά ότι πάντα ε, θα έχω το πνεύμα το συμβιβαστικό, ότι προσπάθησα να εντάξω τις συμβολές όλων ε, σε αυτή την έκθεση και θα ε, λάβω υπόψη μου φυσικά και όλα τα σημερινά σχόλια. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε τον σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ, Κύριε Ματουσέλο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία της και κυρίως επειδή μπόρεσε να μας στέλνει τα έγγραφα όταν τα υποσχέθηκε, πριν δηλαδή τις καλοκαιρινές διακοπές Κάποιες, κάποια βήματα προς την θέση του ΕΛΚ έχουν γίνει, αλλά πρέπει ακόμα να δουλέψουμε έντονα. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα, γιατί το γεγονός ότι οι άνεργοι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να βρουν δουλειά ή να ε, συμπεριληφθούν σε ένα σύστημα είναι κάτι που είναι απαραίτητο πια στην Ένωση. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της δουλειάς μας και γι' αυτό και ζητάμε να παραμείνει στο εσωτερικό αυτό του του προβληματισμού χωρίς να διαχέεται η προσοχή ε, σε διάφορα ε, συστήματα. Οι τροπολογίες μας ακριβώς αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν. Έχουμε ορίσει ότι έχουμε μάλλον ε, συμφωνούμε ότι οι επενδύσει μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση, αλλά κυρίως ότι χρειάζονται διευθυντικές αλλαγές στις αγορές εργασία που θα πρέπει να καταστεί πιο, ε, ε, πιο ελαστική, γιατί το κόστος τη εργασία στην Ένωση είναι απαγορευτικό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία του ανταγωνισμού και τη σημασία των διαγωνισμών. Είναι σαφές ότι χρειάζονται σαφείς κανόνες που να ευνοούν την ε, τον ανταγωνισμό και αυτό επιτρέπει να δημιουργηθεί ένας, μια δυναμική αγορά εργασίας και άρα και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν αποτελεσματικές δομές από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα και από αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Είμαι βέβαιος ότι με την εισηγήτρια θα μπορέσουμε να κάνουμε καλή δουλειά και περιμένω με ανυπομονησία τις επαφές των σκιωδών ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους σοσιαλιστές ο κ. Ιβαν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την συντάκτη για τις προσπάθειές της. Στηρίζουμε ε, την κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η γνωμοδότηση. Το ότι αυξάνονται οι ανισότητε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Οι πλούσιοι γίνονται όλο και πιο πλούσιοι και οι φτωχοί όλο και φτωχότεροι. Υπάρχουν πολλές αιτίε γι' αυτό και νομίζω ότι οι προσπάθειε της Ευρωπαϊκής Ένωση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ε, των παράνομων ροών ε, χρήματος των φορολογικών παραδείσων είναι πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας. Είναι ένας αγώνας τον οποίο πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στους πιο πλούσιους που πληρώνουν τους λιγότερους φόρους. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια σε φορολογικούς παραδείσους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολυεθνικές εταιρείες δεν πληρώνουν ε, φόρους, τους φόρους που πρέπει, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους ε, και ε, ε, αποσύρουν χρήματα, κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις πρακτικές, ώστε οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να στηρίξουν την υγεία, την εκπαίδευση, την, τις υποδομές και να μειώσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, ε, να καταπολεμήσουμε την ανεργία, ώστε να μειώσουμε τις ανισότητες. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συντάκτρια για τις προσπάθειές της και προσβλέπω στι προσεχεί ε, συναντήσει των σκιωδών εισηγητών για να συζητήσουμε περαιτέρω αυτήν την έκθεση. Σα ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Δεν βλέπω κάποιον από το ECR. Καλά τα λέω. Κανείς δεν θέλει. Ναι, καλά, ας μην κάνουμε υποθέσεις τώρα. Λοιπόν, για την Άλντε έχουμε τον κύριο Τρεμόζα που εκπροσωπεί αυτόν. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε την συγγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, αλλά εξ ονόματος ομάδας μου θα ήθελα να πω πως πολλές τροπολογίες των βουλευτών μας ε, θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί υπόψη. Και βεβαίως θα θέλαμε να περιληφθούν κάποιες από αυτές γιατί σε κάποια θέματα έχουμε διαφορετικές απόψεις για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί η ανισότητα. Όπως ξέρετε, στην ομάδα μου υπάρχει μια πλειοψηφία βουλευτών από τις βόρειες χώρες και η αριστερά στη Βόρεια Ευρώπη έχει ένα διαφορετικό όραμα για το τι μπορεί να γίνει για μια κοινωνική Ευρώπη για να μειωθεί η ανισότητα. Είναι πολύ σε συζητήσει αυτές στην ομάδα μας θα θέλαμε λοιπόν ε, να δείτε αν μπορούν να περιληφθούν κάποιες τροπολογίες μας σε κάποιες συμβιβαστικές ε, λύσεις γιατί καθώς δεν είναι δεσμευτικές αυτές οι εκθέσεις αλλά καλό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε συνένεση μεταξύ των ομάδων. Θυμάμαι ότι ήσασταν και πριν από λίγα χρόνια εισηγήτρια για την έκθεση για την ΕΚΤ και έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Για να βρούμε κοινά στοιχεία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Ελπίζω λοιπόν στις επόμενες συνεδριάσεις να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε γιατί θα μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Ίσως λοιπόν να υπάρξει μια συμπερίληψη κάποιων ε, δικών μας προτάσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος, Φίλιπ Λαμπέρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος, όχι από την έκθεση της κυρίας Ματίας, αλλά γιατί χρόνια μετά την έκρηξη του θέματος της, ε, ε, της ε, ανισότητας των ανισοτήτων και μετά από εργασίες πολύ σοβαρές που έχουν επεξεργαστεί τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και ο ΣΑ, όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εδώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουμε ανακοίνωση της Κομισιόν, αλλά για, έχουμε μόνο μια πρωτοβουλία της του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που είναι εντυπωσιακό και μιλώ κυρίως ε, σε αυτούς που επιθυμούν πολύ την ανάπτυξη του ΑΕΠ θα έπρεπε να διαβάσουν την έκθεση του ε, του και του ΣΑ και που λένε όλες αυτές οι εκθέσεις αυτών που είναι ιδιαίτερα ε, φανατικοί οπαδοί της ανάπτυξης ότι όταν υπάρχουν τέτοιες ανισότητες είναι εις βάρος της ανάπτυξης του, της αύξησης του ΑΕΠ. Ίσως λοιπόν γι' αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο στη μείωση των ανισοτήτων, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο θέματα εσόδων ή περιουσίας. Αυτό που διαπιστώνουμε ότι στην κοινωνία μας μπορεί να υπάρχουν ε, και μεγάλε διαφορέ, μεγάλε ανισότητε, όσον αφορά το προσδόκιμο ζωή ε, ανάμεσα στι διάφορε κοινωνικέ ομάδε, Είναι τεράστια διαφορά κάποιε φορέ. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας απασχολήσει αυτό το θέμα, γιατί βέβαια δεν πιστεύω καθόλου πως ε, οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι, όλα τα ανθρώπινα όντα είναι τα ίδια, αλλά... Εδώ πρόκειται για δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν διαπιστώνουμε τέτοιες διαφορές όπως αυτές που επικρατούν σήμερα, Σκεφτόμαστε μια περίοδο ακριβώς πριν από την Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όσον αφορά τη διαφορά τις ανισότητες ε, εισοδημάτων, προσδόκιμου ζωής και ε, ε, ε και διαρωτώμεθα αν ζούμε σε μια δίκαιη κοινωνία. Όπως ε, και για να φέρω το βιβλίο του Μάρτιν Wolf ε, που δημοσιεύθηκε στους ε, The Financial Times, όταν, αν ζούμε δηλαδή σε δημοκρατία, γιατί όταν έχουμε τέτοια ανισότητα ανάμεσα στα έσοδα, είναι, η δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του λαού από τον λαό και για τον λαό, όχι για το 1 ή το 2 ή το 3% του λαού. Είναι δύσκολο να στηρίξουμε ότι ασκούμε πολιτικές δημοκρατικού τύπου όταν από αυτές ωφελούνται, όπως το διαπιστώνουμε από την κρίση και έπειτα, ότι αυτές ωφελούν μια μικροσκοπική πλειοψηφία. Και αυτό να το πω και στον κύριο Μαρτουτσέλο, ο οποίος μας έκανε την τιμή να φύγει μόλις έκανε αυτή την παρέμβαση, που πραγματικά Απορώ και εξίσταμε όταν ε, ακούγονται τέτοια πράγματα ώστε να μειωθούν, για να μειωθούν οι ανισότητες, όπως αυτά που είπε ο κ. Μαρτοτσέλο, ότι δηλαδή πρέπει να μεταρρυθμιστεί η αγορά της εργασίας για να μειωθούν οι ανισότητες. Μα δεν είναι οι ανισότητες ε, δεν οφείλονται στην ατμοσφαιρική πίεση ή στην κλιματική αλλαγή. Εδώ και 30 χρόνια αυξάνονται οι ανισότητες. Υπήρξε μια πολιτική καμπή και μια πορεία που ακολουθήθηκε. Και αυτή η καμπή είναι η αποδυνάμωση όλων των συστημάτων κοινωνική αλληλεγγύη στα κράτη. Πρόκειται για αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για αποδυνάμωση της ε, ε, διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων υπέρ της ε, ισχύω, της αύξησης της ισχύω ε, ε, του κεφαλαίου. Αυτό είναι η κοινωνική ε, παρουσία. Να θυμίσω τον κύριο Μαρτουτσέλο που είναι και Ιταλός μάλιστα ότι το ποσοστό απασχόληση είναι στα 50%. Πώς βρίσκει κανείς φουλ δουλειά σε μια χώρα μέσω διορθωτικών αλλαγών, μόνο δηλαδή αν μειωθούν οι ακαμψίες της αγοράς εργασίας. Όταν δεν υπάρχει καμιά ανάπτυξη και ελαστικότητα, δεν θα δεν πρόκειται να υπάρξει απασχόληση στην Ιταλία. Θα πρέπει να προβλεφθούν και άλλες μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στο να ζουν όλοι μια αξιοπρεπή ζωή. Η νέα γενιά στην Ιταλία, η νέα γενιά στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης de facto δεν μπορεί να πιστέψει πια στην υπόσχεση μιας, αξιο... μιας αξιοπρεπούς και βιώσιμης και διαρκούς εργασίας. Και όταν βλέπουμε μηδενικά συμβάσεις μηδενικών ορών αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνο κατόνομα εργαζόμενοι και στην πραγματικότητα είναι φτωχοί είναι τελείως πρόσχερη η δουλειά τους και ζουν σε αναξιοπρεπείς συνθήκες. Καταλαβαίνω αυτό που λέει και ο συνάδελφος Τρεμόζα, ότι πρέπει να καταλάβουμε τα όσα είναι ενδιαφέροντα από τις προτάσεις του Ισάλντε. Να κλείσω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναθέσει το θέμα της δικαιοσύνης και άρα της μείωση των ανισοτήτων στην καρδιά των πολιτικών, των δημόσιων πολιτικών, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Εξαμήνου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κάποιοι συνάδελφοι δεν μίλησαν. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιον λόγο στο Catch Να δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια πάλι για να συνοψίσει. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα απαντήσω στους συναδέλφους που είναι εδώ. Είχαμε και μία συνεδρίαση των σκιωδών ε, την Δετάρτη. και την, τετά... Μάλλον θα έχουμε συνεδρίαση, με συγχωρείτε, και θα έχουμε έτσι και την ευκαιρία να συζητήσουμε σε με λεπτομέρειε όλα αυτά τα θέματα, αλλά προφανώ έχω να πω ε, πράγματα στου συναδέλφου του ΕΛΚΑ και των Σοσιαλιστών, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το χρόνο να απαντήσω, γιατί θα έχουμε την Τετάρτη τη δυνατότητα να το κάνουμε. Σε όσα είπε τώρα ο Ραμών και το θέμα των τροπολογιών των φιλελευθέρων. Πρώτον, Όλες οι τροπολογίες δεν έχουν περιληφθεί στις συμβεβαστικέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τις μελέτησα. Τις μελέτησα, αλλά καλύτερα θα είναι να ψηφιστούν χωριστά, γιατί είναι παράγραφες αυτές καθεαυτές και αφορούν θέματα διαφορετικά από τις υπόλοιπες τροπολογίες. και άλλες δεν τις έλαβα υπόψη γιατί είναι τελείως ε, αντίθετες με ε, τα όσα πιστεύω ότι θα αποτελέσουν μια λογική συμβαστική λύση για αυτή την έκθεση. Δεν ε, το έκανα μόνο για τροπολογίες δικές σας των φιλελευθέρων, αλλά και για άλλες που ήταν δύσκολο να ενταχθούν σε συμβαστικές. Αλλά μέχρι την Τετάρτη θα δούμε, θα μπορέσουμε και να τα συζητήσουμε ε, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε. Για τα σχόλια του Φιλίπ ε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι πρέπει να συζητήσουμε και συζητάμε αυτά τα θέματα εδώ και τόσα χρόνια. Είναι πραγματικά γελίο το να πρέπει να κάνουμε απλά μια έκθεση πρωτοβουλία εμεί, αλλά γι' αυτό ακριβώ και πιστεύω πω είναι ακόμα περισσότερο ένας λόγος για να ε, κάνουμε αυτή την έκθεση, να, ε, να μιλήσουμε εμεί ω κοινοβούλιο. Σε πολλού τομεί δεν έχουν, έχει γίνει τίποτα λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ε, αναζητήσουμε συμβιβαστικέ και για αυτά τα ζητήματα. Το θέμα της δικαιοσύνης αλλά και της δημοκρατίας θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Αν έχετε και άλλα θέματα μέχρι Τετάρτη, παρακαλώ να μου τα στείλετε. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε όλα τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Thank you, Maria. This is... Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώνουμε την σημερινή συνεδρίαση ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 25 Σεπτεμβρίου, στην ΕΜΠΛ τρεις μέρες μετά, 28 Σεπτεμβρίου, και στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώσαμε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Δεν έχουμε κανένα θέμα στα διάφορα από ό,τι γνωρίζω και η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, 3 ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.